εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ευρωπαϊκά χρήματα Έχουμε την ε, κατάρτιση και τον εξοπλισμό συνεροφυλάκων στον Ήγυρα για να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και να συλλαμβάνουν μετανάστες. Όμως τώρα η συνέπεια είναι ότι άλλοτε σίγουρα οδοί μετανάστευσης ε, τώρα είναι ο επικίνδυνο οδείο που έχουμε απαγωγές ε, και παραβιάσεις. Και οι πολιτικές σας φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί από τις ίδιες τις μαφίες. Θα συνεχίσουμε να μεταναστεύουμε σε έλεγαν άνθρωποι από το Σουδάν, άνθρωποι που είχαν δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώ του συνέλαβαν και του βασάνισαν στη Λιβύη. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό, κύριος Λεμπρετό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω ο ΙΕ με το σύμφωνο του Μαρακέ, η Επιτροπή των Βρυξελών πιστεύει ότι το φαινόμενο τη μετανάστευση που είναι κατακλυσμιαίο είναι κάτι το αναπόφευκτο που το δεχτούμε ω πεπρωμένο. Με τρία παράλογα μέτρα προσπαθεί να το επιλύσει. Την έγκριση του τέταρτου κανονισμού του Δουβλίνου που θα κατανέμει του ε, μετανάστε μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών ε, μέσω υποχρεωτικών ποσοστώσεων. Δύο. Η νόμη μεσοδή μετανάστευση. Τρία. Η εγκατάλειψη των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Κάτι που πολλά ευρωπαϊκά κράτη όμω έχουν επαναφέρει εδώ και δύο χρόνια, αντιδρώντα στο παράλογη συμφωνία του Σέγγεν. Κανένα, κανένα από αυτά τα τρία μέτρα δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Θα καταλήξουν σε αποτυχία όπω το πρόγραμμα Juncker το 2015 που σκοπό είχε να εγκαταστήσει 160.000 μετανάστε και στο οποίο αντιστάθηκαν δικαίω πολλά ευρωπαϊκά κράτη για να διαφυλάξουν την εθνική του ταυτότητα. Οι ευρωπαϊκοί λαοί είναι θνητοί. Το ξέρουν και δεν θέλουν να φανιστούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι και εκείνη θνητή αλλά φαίνεται να το αγνοεί. Δεν ακούει τη φωνή των ευρωπαϊκών λαών. Εκείνη λοιπόν θα χαθεί. Για 1,5 ναι. λεπτό, για 1,5 λεπτό Σκοέλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Βραμόπουλε, κυρία Υπουργέ τις πρώτες δύο εβδομάδες της νέας χρονιάς ένας άνθρωπος τη μέρα πέθαινε προσπαθώντας να φτάσει τα σύνορά μας. Πέρσι, το 2018, είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό ε, θανάτων, έναν νεκρό ανακατό αφήξης. Όλο ένα λιγότερε οι αιτήσει για άσυλο. Εν τω μεταξύ όμω, πέντε χώρε συνεχίζουν να υποδέχονται περίπου 75% των ε, αφιχθέντων. Ξέρουμε τι λένε οι λέκιστες ε, τα τελευταία χρόνια ε, και ξέρουμε ότι μερικές φορές ε, λένε ότι όσοι δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Ευρώπη επιστρέφουν στους χώρους τους και αυτό είναι σωστό. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Οι κυβερνήσεις έχουν υπολείπονται το καθηκόν του μάλλον. Ε, το 2017 η αποτελεσματικότητα των ε, επιστροφών έφτασε το 37%, το χαμηλότερο ποσοστό από τα προηγούμενα χρόνια. Θα πρέπει να ενισχύσουμε, μάλλον μπορέσαμε να ενισχύσουμε την ε, Frontex και θέλουμε να το ξανακάνουμε με ένα σύστημα ασύλου και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό γι' αυτό, με οκτώ δομικά μέτρα που τα ανέφερε και ο κύριος Ντεμέρα. Όμως δεν θα πετύχουν αν δεν δράσουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Γι' αυτό κύριε Υπουργέ θα μας ακούσετε ποτέ στο Συμβούλιο, από το Κοινοβούλιο, θα κάνετε κάτι στους τέσσερι μήνε της Προεδρίας σας. Δεν μπορούμε απλώς να προστατεύουμε την επικρατειά μας, διότι αυτό ε, θέτει να αμφιβόλω την εικόνα μας στον υπόλοιπο κόσμο. Κάνει ε, αδύναμο, το σεβασμό προς τις αξίες μας και ουσιαστικά ενθαρρύνει τους εθνικισμούς, τους εγωισμούς και το λεκισμό χωρί νόημα. Σα ευχαριστούμε για ένα λεπτό, κύριο Νίντερ Ευχαριστώ ε, όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες. Η Λένδη και τα σκάφη γεμάτες μετανάστες, γεμάτες που φτάνουν στην ε, Μεσόγειο, μας έχουν φέρει στην σημερινή κατάσταση. Ένα μέρος των κρατών μελών με την υποκριτική τους στάση δεν θέλουν να υπογράψουν ε, την αναθεωρημένη εκδοχή, την ένταρτη εκδοχή του κανονισμού του Δουβλίνου. Και το Συμβούλιο δεν φαίνεται να μπορεί να αναλάβει το ρόλο που του αναλογεί. Ε, χρειάζεται ένας νέος κανονισμός του Δουβλίνου, είναι σαφές. Χρειάζεται νέα προσωρινή συμφωνία μέχρι να γίνει αυτό και ε, μέχρι να αναλάβουν οι επόμενοι στη νέα θητεία θα πρέπει να διαφυλάξουμε την προστασία των μεταναστών που φτάνουν στην Ευρώπη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι πρόθυμα, ιδάλλως να πληρώσουν, να πληρώσουν ε, ε, μια ποσόστοση. Κυρία ε, Υπουργέ, κύριε, ε, θα πρέπει το Συμβούλιο να σκεφτεί την προσωρινή εφαρμογή μέτρων, ιδάλω δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ήθελα να ακούσω το τέλο τη παρέμβασή σα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Βίστησεν για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κάθε χρόνο έχουμε πολλούς λαθρομετανάστες που περνούν τα ευρωπαϊκά σύνορα. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δίνει την εντύπωση ότι υποστηρίζει τους εμπόρους και τους λαθρομετανάστες χωρί να βοηθά του νόμιμους μετανάστε που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Και πολλοί ευρωβουλευτέ φαίνεται να πιστεύουν ότι αν νομιμοποιήσουμε το καθεστώ των ε, εκατομμυρίων ανθρώπων αυτών που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη χωρί ε, καμία προπόθεση, κανέναν όρο, θα πάνε όλα καλά. Από την πλευρά της Δανίας όμως ε, το σημαντικό ε, είναι ότι θέλουμε κάποιοι να έρθουν αλλά όχι Ατάκτος, το μόνο ε, θεσμικό όργανο που ανέλαβε κάποιο μέτρο εδώ ήταν το Συμβούλιο που αντιστάθηκε και είπε όχι, όχι στην ομορμοποίηση της λαθρομετανάστευσης όπως την προτείνουν το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σοβαροί και σοβαρά ε, ε εκπροσωπούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση πριν φτάσουν όλοι αυτές στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε κυρία Αλμπιόλ Γκούσμα. Καταρχήν, ε, αποφασίσατε να κλείσετε τα σύνορα προκειμένου κανένα μετανάστε να μην πατήσει πόδι στην Ευρώπη. Μετά, αποφάσισαν ότι η καλύτερη στρατηγική αποτροπή είναι να του αφήνουμε να πεθαίνουν ε, στην ε, Μεσόγειο και αφήνονται στα χέρια τη μαφία. Δεν έχουμε εδώ πλοία που να χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή ούτε επιτρέπεται στι ΜΚΟ να σώζουν ζωέ. Και η κυβέρνηση τη της ε, Ισπανίας επιτρέπει στο Περνέλη να σώσει ε, ανθρώπους ε, και και τελικά μετατρέπεται και αυτή σε δολοφόνο. Έχουμε τώρα το νέο, τη νέα πικιοκρατία και υλοποιείται με συμφωνίες με τις αφρικανικές χώρες όπου με ευρωπαϊκά χρήματα χρηματοδοτούνται κέντρα βασανισμών τα ε, κονδύλια ε, στέλνονται στην Αφρική και φτάνει σε συμφωνίες ε, με δικτάτορες η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως με το Σουδάν και τελικά βλέπουμε έναν λόγο που αναπτύσσεται από την ακροδεξιά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σεζάμι Τιμέχ για ένα μισή λεπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Όταν ε, αναφερόμαστε στα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας, όταν δηλαδή είχαμε ανθρώπους οι οποίοι υπέφεραν επί τρεις ε, εβδομάδες, 49 άτομα, κατάφεραν να αποβιβαστούν και επιλύθηκε επιτέλους αυτό το θέμα επιλύθηκε με τρόπο διαχείρισης κρίσεων με συνεννοήσεις μεταξύ πρωθυπουργών και ο Πρωθυπουργός και ο, και ο Επίτροπος και εξέφρασε ένα συνέστημα ευρωπαϊκό όταν είπε ότι αυτό θα έπρεπε να εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί στην πραγματικότητα θέλουμε έναν βιώσιμο μηχανισμό που θα βασίζεται στις δικές μας αξίες της αλληλεγγύης και να μην ε, το αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση. Έχω και κάποια άλλα σχόλια. Ασκείται πίεση και εκφοβισμός από τις μεγάλες χώρες στις μικρές. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Και επίσης ε, πρέπει να δούμε το ζήτημα. Υπάρχει μια σαφής ε, πολιτική επιστροφών αυτό θα ισχύει για όσους ε, δεν έχουν δικαίωμα να έρθουν στις ε, χώρες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τα σχόλιά του για τη Μάλτα και είπε ότι θα επανέλθει στη Μάλτα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει έρθει και τον ε, περιμένουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Μωραή για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πλησιάζουμε το τέλος της έντολής μας. Έχουμε ένα παραθύρο τριών μηνών μόλις και κάπου τα έχουμε ξαναδεί όλα αυτά. Μια μικρή χώρα όπως η Μάλτα, 400.000 ανθρώπων, όταν πρώτο έγινα ευρωβουλευτής ε, δεχόταν πρόσφυγες και πάλι η χώρα αυτή δέχεται πρόσφυγες και πάλι ε, περιφέρεται από κράτος μέλος ε, σε κράτος μέλος ο Επίτροπος αναζητώντας λύση και πάλι λέμε ότι δεν έχουμε κάποια λύση και κάποιο πακέτο. Αυτή την ερώτηση πρέπει να απαντήσουμε και η απάντηση είναι ότι χρειάζεται κάποια κοινή προσέγγιση. Αλλιώς ε, το έσχος του Sea-Watch θα επαναληφθεί, πάνω από 2.000 άτομα θα πεθάνουν ε, και θα αυξηθούν οι αριθμοί. Έχουμε λοιπόν ε, τρεις μήνες ένα παράθυρο ευκαιρίας δεν είχαμε την ειδική πλειοψηφία επί Αυστριακής Προεδρίας και ζητώ από την Ρουμανική Προεδρία να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία. Πρέπει να έχουμε ειδική πλειοψηφία με τις συνθήκες, πρέπει να γίνει κάτι. Πολλοί από τους ηγητές ήταν εδώ στο Κοινοβούλιο. Να εκμεταλλευτούμε, κύριε Πρόεδρε, την ευκαιρία. Έχουμε τρεις μήνες. Σας ευχαριστώ. Ράντεφ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, μιλάμε για την κρίση στη Μεσόγειο. Δεν υπάρχει όμως μια κρίση αυτή τη στιγμή, ούτε τεράστια αριθμή. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κολλήσει για το που θα πάνε 40 άτομα. Και αυτό μετά την αποτυχία της να μετακινήσει χιλιάδες ανθρώπους από την Ιταλία και την Ελλάδα και αφού απέτυχε να μεταρρυθμίσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και Μετανάστευσης. Κυρίες και κύριοι, ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές μεταναστευτικές κρίσεις είναι να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του ασύλου για να είναι σαφές το ποιος είναι υπεύθυνο για τους ετούντε άσυλο, ποιος ε, εξετάζει τις αιτήσει ε, και πόσο διακρίνουμε μεταξύ ετούντων των και οικονομικών μεταναστών. Ε, πρέπει ακριβώς να ελαφρυνθούν οι χώρες πρώτης γραμμής, η Μάλτα, Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία. Ε, είμαι σίγουρος ότι όλα τα κρατημέλη, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται στον χάρτη, θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό και ο Αγαπητοί ε, συνάδελφοι, πριν από λίγες ημέρες είδαμε το κοινικό παιχνίδι με 49 ανθρώπους που έσωσαν η Μίκιο και επιτέλους ε, τελείωσε. Τα πλοία μετά από 18 ημέρες ε, έφτασαν με ανθρώπους με ψυχικά τραύματα. Ε, προσεχώς θα τεθεί ξανά το ερώτημα ποιος θα προσφέρει ασφαλή λιμένα στα πλοία και θα μοιραστούν οι διασωθέντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτύχουν πάλι τα κρατη Και αυτό χρειάζεται αμέσως μια λύση. Πρέπει να υπάρξει ένα συνασπισμό των προθήμων κρατών μελών με μια μόνιμη κλίδα κατανομής και εξακολουθεί το Συμβούλιο να αρνείται να διαπραγματευτεί σοβαρά. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ακριβώς περιέχει αυτήν την αλληλεγγύη για την οποία συνεχώς μιλάμε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ε, επιτέλους ε, να φτιάξει ένα δικό της πρόγραμμα διάσωσης για να σταματήσουν οι θάνατοι Μεσόγειο. Σας ευχαριστώ. Μάντλ για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι σχεδόν πουθενά αλλού στον ε, κόσμο δεν ε, ζουν έτσι τις αξίες του ανθρωπισμού όπως στην Ευρώπη. Και αυτό οδηγεί και στην ευημερία της Ευρώπης και την κάνει τόσο ελκυστική. Αυτό αποτελεί και μια ευθύνη της Ευρώπης για μια ισχυρή Ευρώπη με αυτές τις αξίες και για τους ανθρώπους που κινδυνεύουν. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα σύστημα το οποίο θα βοηθάει πραγματικά αυτούς οι οποίοι το χρειάζονται και όχι εγκληματικές συμμορίες διακινητών. Δεν υπάρχει κρίση, όπως λέει ο κύριος ο Επίτροπος. Αυτό οφείλεται στο ότι σταμάτησε η εγκληματική διακίνηση μέσω της Μεσογείου και των Βαλκανίων. Με αυτό δεν έχουν μειωθεί οι θάνατοι. Πρέπει να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα και κυρίως να ασχοληθούμε με την ένταξη στην Ευρώπη για τους ασθενέστερους. Πώς χρειαζόμαστε κιόλας. Η κυρία Κιέγγε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εδώ και πάνω από ένα χρόνο το Κοινοβούλιο ψήφισε τη μεταρρυθμίση του κανονισμού του Δουβλίνου, μία καινοτόμο ε, μεταρρύθμιση που επικεντρώνεται στην αρχή της αλληλεγγύης. Χωρίς αυτή τη μεταρρύθμιση δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι δυνατό να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό φαινόμενο χωρίς ε, σαφή καθορισμό των ευθυνών και χωρίς καμία εγγύηση της προστασίας των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών ε, ντροπιαστική υπόθεση του Aquarius και του Sea Watch ε, θα γίνουν πρακτική. Ευχαριστώ όλε τι ΜΚΟ που ανέλαβαν ε, την έρευνα και τη διάσωση. Θα πρέπει να ανακτήσουμε την ανθρωπιά μα. Καταρχήν, να σώζουμε τι ανθρώπινε ζωέ. Θα πρέπει να του ε, σώσουμε και να του οδηγούμε στον πρώτο ασφαλέ λιμάνι. Και θα πρέπει να ζητήσουμε δικαίωμα σε άμεσο ελιμενισμό των σκαφών. Επίση, θα πρέπει να υπάρχει επιμερισμό των ευθυνών ευθυνών. Υπάρχουν ε, διάφορες, ε, στις διάφορες κυβερνήσεις ζητώ να εγκαταλείψουν τη δημαγωγία και να αποφασίσουν ε, σύμφωνα με τις συνθήκες αλλά και σύμφωνα με τα δύο σύμφωνα που υιοθετήθηκαν πρόσφατα από τα Ηνωμένα Έθνη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω πολλούς ομιλητές για το ΚΑΤΣΔΙ. Θα βάλω τα δυνατά μου να τους δώσω το λόγο. Ο κύριος Αγγιλάρ καταρχήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπουμε δυστυχώς με θλίψη αυτή την νιωστή συζήτηση για το εργοδοστευτικό και ε, εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναρωτιούνται και στρέφονται προς το Συμβούλιο και τους ρωτούν τι πίστευαν οι προκατοχοί σας όταν ε, υπέγραψαν τη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, που υποσχόταν ακριβώς αυτό που υιοθέτησε ως θέση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκφράσαμε τη θλίψη μας επειδή δεν έγινε σεβαστή αλληλεγγύη, ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα σύστημα επιμερισμού της ευθύνη στη διαχείριση των αιτήσεων ασύλου πρέπει να αναλυφθούν οι ευθύνες από το Συμβούλιο, γιατί θέλουμε μια αποτελεσματική ανθρωπιστική ευρωπαϊκή πολιτική. Και οι ευθύνε του Συμβουλίου δεν λύνονται ούτε ε, με έκτακτα μέσα, ούτε με τηλεφωνικές κλήσεις, ούτε ποινικοποιώντα τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Συγγνώμη, έλειξε ο χρόνο σα, λέει πρόεδρο. Κυρία Τόμαση, θα είμαι πολύ αυστηρή για το ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια κράτη-μέλη συμμετείχαν πολύ ευχαριστώ σε κάποιες επεμβάσεις στα αφρικανικά κράτη και μιλούσαν για δημοκρατία. Τώρα πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν, έχουν διαλυθεί αυτά τα αφρικανικά κράτη δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κάποια από αυτά για να σταματήσουμε τις μεταναστευτικές ροές. Αυτό σημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να προστατεύσει τα εξωτερικά της ε, σύνορα και να σταματήσει την ε, παράνομη διακίνηση και να υπάρξει μια έφτακτη πολιτική μεταναστευσής. Ε, και για να λειτουργεί ακριβώς αυτή η πολιτική πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός ε, οικονομικών μεταναστών, ε, μεταναστών και πραγματικών προσφύγων. Αυτό ακριβώς είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Κύρια Πρόεδρε, κύριε Επιτροπή, το 2019 σημαντικό έτος. Πρέπει να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα Γι' αυτό ζητάμε εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματική πολιτική ε, μετανάστευσης. Και κύρια Στίβενς, εμείς και ο κύριος Φερχόφστατ δεν ζητάμε ανοιχτά σύνορα. Θέλουμε να μην διαλέγουν πού θα πάνε οι ε, πρόσφυγες, ε, να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των κατών μελών, να προστατεύουμε τα παιδιά και να αντιμετωπίσουμε τους ε, λαθροδιακίνητες, να μεταρρυθμίσουμε το Δουβλίνο και αναγνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν μόνο τους, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και υπάρχουν κάποιοι που διακινούν ε, ψεύτικους αριθμούς, θα πρέπει να ντρέπονται. Ερωτώ Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Πρέπει επιτέλους να κάνουμε κάτι, να περάσει τώρα το πακέτο. Ευχαριστώ κύριο Σολέ. Ευχαριστώ. Η αντιευρωπαϊκή ακροδεξιά κερδίζει έδαφο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν διάφορε κριτικέ για να αντιμετωπίσουμε αυτό. Μία από την Ανδαλουσία ε, ουσιαστικά ε, με μέλη του ε, Λαϊκού Κόμματο προσπαθεί να απομονώσει την δεξιά. Το άλλο είναι αυτό που συνέβη στη Σουηδία, απομόνωση τη ακροδεξιά. Και Επίσης, το πιο κοινό ε, που κάνουμε είναι να υιοθετούμε τις απλουικές συνταγές της ακροδεξιάς, κυρίως σε θέματα μετανάστευσης. Ε, με αυτόν τον τρόπο εξηγείται, τουλάχιστον εν μέρη, ότι χρόνια μιλάμε για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, ότι χρόνια μιλάμε για τη μεταρρύθμιση του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου και τα κράτη-μέλη είναι ανίκανα να συμφωνήσουν ε, δείχνοντας ε, μία τεράστια έλλειψη αλληλεγγύης και βούλησης επιμερισμού των ευθυνών ε, και να εκχωρήσουν κυριαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εγκαταλείψετε τους εγωισμούς και τον λογικισμό και να ελοπίσουμε αυτή τη μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ κυρία Κούνεβα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα της μεταναστευτικής κρίσης, μαλώνουμε ακόμα για το πόσους πρόσφυγες και μετανάστε θα δεχτεί κάθε κράτο το έδαφο του όχι για να του κάνει πολίτε του, αλλά να εξετάσει αν δικαιούνται άσυλο. Είναι ντροπή για την Προεδρία και το Συμβούλιο να μας λέει πώς το πρόβλημα είναι οι δευτερογενείς ροές και πώς η αλληλεγγύη δεν είναι το μοίρασμα των απελπισμένων ανθρώπων. Τι είναι αλληλεγγύη κυρία Προεδρεύουσα, να δίνονται χρήματα για να χτίζουμε καταβλισμούς, οι δευτερογενείς ροές θα υπάρχουν όσο είναι κλειστή η πόρτα και δεν σταματήσουμε τους πολέμους. Είναι πολύ άσχημο να ακούγεται η φράση παράνομοι πρόσφυγες και μετανάστες. Οι άνθρωποι δεν μπορεί να είναι παράνομοι. Παράνομος είναι ο πόλεμος και παράνομο είναι το εμπόριο όπλων και εμείς αυτά δεν τα συζητάμε καν πόσο ακόμα παιδιά και γυναίκε πρέπει να φύγουν από τη ζωή να σταματήσουμε του πολέμου. Ευχαριστώ. Thank you, colleagues. Uh, taken five... ευχαριστώ. Ακούσαμε πέντε παρεμβάσεις στο Catch the Eye. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους υπολείπους. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον Επίτροπο να απαντήσει στην συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπο. Ναι, πριν μιλήσετε, πράγματι ήσασταν από τις ε, πρώτες, αλλά ε, λυπούμε. Ειλικρινά αν ήταν δική μου η απόφαση θα σας έδινα περισσότερο χρόνο, αλλά ήδη ε, υπάρχει πίεση από τους ανωτέρους μου. Κύριε Αμπραμόπουλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ επίκαιρη συζήτηση. Θα ευχόμουν να μην τη χρειαζόμασταν, αλλά δυστυχώς τη χρειαζόμαστε. Όπως ε, είπα νωρίτερα και όπως πολλοί από εσά ε, τονίσατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία της Ευρώπης. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ προσωπικά αναλαμβάνουμε πλήρη δέσμευση να συνεχίσουμε να συνεργαστόμαστε μαζί σας και με το Συμβούλιο για να πετύχουμε αυτό τον πολύ σημαντικό στόχο, τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ξεκάθαρη και ηχηρή υποστήριξη. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εντατικά για να πετύχουμε την ολοκλήρωση του συνολικού μας έργου και για να απαντήσω στην κυρία Ιντβελτ, Σοφή, όλες οι προτάσεις μας είναι απαραίτητα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης πολιτικής. Σημείωσα τις παρατηρήσεις σου και ξέρω πόσο σε απασχολεί το θέμα και το σέβομαι, αλλά από τη δική μας σκοπιά εμείς έτσι βλέπουμε το όλο πακέτο και την πολιτική που πρέπει να υιοθετήσουμε. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στον τομέα της μετανάστευσης όλες μας οι δράσεις αλληλοσυνδέονται και θα πρέπει όλα τα κομμάτια να ταιριάξουν μεταξύ τους. Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης για το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια απαραίτητη μεταρρύθμιση για να καταπολεμήσουμε την παράτυπη μετανάστευση, να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τις δευτερογενείς μετακινήσεις και να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ταχεία εξέταση των αιτήσεων ασύλου σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι η συνεργασία με τις τρίτες χώρες είναι κλειδί, όχι μόνο για να ε, εμποδίσουμε τις παράνομες αναχωρήσεις για την Ευρώπη, αλλά και για να μπορέσουμε να δώσουμε τέλος ε, στην ε, δράση των διακινητών και των λαθρεμπόρων. Η αυξημένη συνεργασία με τις ε, χώρες εταίρους από την Αφρική είναι μέρος της σκληρή μας δουλειά. Ε, το καταπιστευτικό ταμείο για την Αφρική έχει παρουσιάσει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Επίσης, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παράκτια κράτη στη Μεσόγειο θα είναι έτοιμα και ικανά να υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου ό,τι αφορά την έρευνα και τη διάσωση. Ένα ζωτικό στοιχείο, επομένως, είναι και η δική μας δουλειά για τις επιστροφές και με τις χώρες προέλευσης, αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις δράσεις μας για να ενδυναμώσουμε και να διαχειριστούμε καλύτερα τα κοινά εξωτερικά μας σύνορα. Η πρότασή μας για ένα μόνιμο σώμο 10.000 συνοριοφυλάκων είναι επιτάπητος. Αυτό ζήτησαν τα κράτη-μέλη και εμείς το παραδώσαμε. Γι' αυτό πρέπει επίσης να προωθήσουμε τις προτάσεις αυτές και είμαστε σχεδόν έτοιμοι ή έτοιμοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον. Ένα απρόβλεπτο μέλλον. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων. Δεν μπορούμε πλέον να έχουμε τέτοιες ανοργάνωτες λύσεις ad hoc. Τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να μετατρέψουμε τα λόγια σε πράξεις. Σε αυτό το εκλεγικό νέο έτος θέλω να επαναλάβω το μήνυμα ότι η Ευρώπη θα κρυθεί από τα αποτελέσματα που παρουσιάζει στους πολίτες, όπως είπε και η Σεσίλια. Οι πολίτες μας περιμένουν πολλά από εμά και βασίζονται σε εμά. Ελπίζω σύντομα να έχουμε μια διαφορετική συζήτηση και να συζητήσουμε κυρίως νομοθετικούς φακέλους. Ας προχωρήσουμε λοιπόν και θα πρέπει να είναι ο στόχος μας μια ισχυρή κληρονομιά για το μέλλον της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επιτροπή. Να δώσω τώρα το λόγο στην Υπουργό Εξωτερικών, κυρία Τσιώτη, για το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση που σήμερα συζητήσαμε είναι πραγματικά ατυχή. Η Προεδρία εργάζεται άκουνα σε συνεργασία με την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη για να καταλήξουν σε, μια, σε έναν κανονισμό που να επιτρέπει προβλεψιμότητα και να συμφωνεί με το Διεθνέ Δίκαιο τη Θάλασσα για την ε, ε, επαναγκατάσταση και τις αποτελεσματικές ε, υποβολές αιτήσεων ασύλου και τον Δεκέμβριο του 2018 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο να συνεχίσει τις προσπάθειές του βάσει των προηγούμενων συμπερασμάτων του, τα οποία θέλω εδώ να παραθέσω να αναζητήσει συνένεση για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου βάσει μια σωστά εξισορροπημένη κατανομή ευθυνών και έκφραση αλληλεγγύη. Λαμβάνοντα υπόψη ότι οι αποβιβάσει ε, μετά τη διάσωση στη θάλασσα είναι γεγονό. Η Ρουμανική Προεδρία θα αναλάβει λοιπόν τι ευθύνε τη ε, βάσει αυτή τη κατεύθυνση. Σε πολυάριθμε περασμένε προεδρίε έγιναν ε, αμέτρητε προσπάθειε για να βρεθεί μια λύση αποδεκτή από όλου. Διαφορετικέ ε, συνταγέ δοκιμάστηκαν, όμω μέχρι τώρα δεν υπήρξε συμφωνία. Δεν υπήρξε καμία συμβαστική λύση που να ικανοποιεί όλου. Όπω λοιπόν έγινε σαφέ, οι συμφωνίε θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τι διαφορετικέ πτυχέ μια σφαιρική προσέγγιση. Αυτή είναι και η ε, οδό που θέλει να ακολουθήσει η Ρουμανική Προεδρία. Όπω προείπα, εργαζόμαστε για να βρούμε μια διευθέτηση που να επιτρέπει να υπάρξει προβλεψιμότητα και ε, συνέπεια με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Οι αποβεβάσεις να είναι εφικτές και ε, το σύστημα ασύλου αποτελεσματικό. Η λύση που βρέθηκε την, ε, την προηγούμενη εβδομάδα για τα δύο σκάφη ανθρωπιστική βοήθειας είναι ευπρόσδεκτη και σωστά υποστήριξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και την ΕΑΣΟ την εξέβρεση αυτή τη λύση. Είναι ύψη τη σημασία να πετύχουμε γρήγορα το στόχο μα. Ε, έστω ε, και με μια προσωρινή λύση που όμω θα πρέπει να γίνει μόνιμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι και οι μετανάστε οι ίδιοι δεν αξίζουν η κατάσταση αυτή να παραμένει ανεπίλητη. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη μεταρρύθμιση των κοινών κανόνων ασύλου κάτι που θα επιτρέψει μια λύση διαρκεία, μια μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και στο μέλλον. Παραμένω πεπισμένη ότι χάρη στι προσπάθειε όλων μα μπορούμε να ε, διαδραματίσουμε ένα σοβαρό βήμα προόδου προ την επιτεύξη του στόχου μα. Και πάλι σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και για τη συνεργασία σας κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής συζήτησης. Τώρα λίγη συζήτηση. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει δηλώσει του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επισκόπηση τη Αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου. Να θυμίσω σε όλου του συναδελφού ότι για τη συζήτηση αυτή προβλέπεται διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ, Δεν προβλέπεται μόνο διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ και δεν θα γίνουν δεκτέ και ε, δεκτά αιτήματα γαλάζια κάρτα. Πριν δώσω το λόγο στον κακελάριο Σεμπάστιαν κουρτ, να ευχαριστήσω την Αυστριακή Προεδρία για την εντατική συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο. Θα ευχαριστήσω επίσης την Αυστριακή Προεδρία για την πρόσκληση προς το Ευρωκοινοβούλιο να συμμετάσχει στην ε, εκδήλωση για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική, τη Σχετική Σύνοδο, όπου συμμετείχαν και ο πρόεδρος, ο Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούνκερ, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Τούσκ, και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η όλη σύνοδο. Ευχαριστώ του εκπροσώπου και τη αυστριακή κυβέρνηση που συμμετείχαν στι ε, συνόδους του Κοινοβουλίου και σας ευχαριστούμε και για την έλευσή σα στι Βρυξέλλε. Με όλε αυτέ τι ευχαριστίε, δίνω το λόγο στον καγκελάριο Κούρτ. Κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν, κύριες και κύριοι πρόεδροι των ομάδων και βουλευτές. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της Αυστριακής Προεδρίας. Έχουμε πίσω μας έξι εντατικούς μήνες, ένα πολύ πυκνό πρόγραμμα εργασίας και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα ευθύς ξερχής να αναφέρω την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιών. Και σας ευχαριστώ για την στήριξη στην Προεδρία μας. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, πάντα αποδίδω μεγάλη σημασία στην συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Μπόγνερ Στράου ε, και την Καρολίνα Ερστάτλερ, τις υπουργού που μας εκπροσώπησαν στις ημέρες της Ολομέλειας. Θα ήθελα όμως να σας ευχαριστήσω και για τους 161, ε, τις 161 συναντήσεις στα πλαίσια του διαλόγου που είχαμε. Να ευχαριστήσω λοιπόν Συμβούλιο Κοινοβουλίου και Κομισιόν για την διάθεση συμβιβασμού που επέδειξαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα της Αυστριακής Προεδρίας, ε, τον πρέσβηρά μας, ε, τον Αλεξάνδρ Σάινμπεργκ και τους άλλους της ε, Βρυξέλλες. Και βεβαίως επειδή κάθε προεδρία είναι μόνο ένας κρίκος στην αλυσίδα, να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους στο τρίο, την Εστονία και την Βουλγαρία. Και δράτουμε της ευκαιρίας ε, για να ευχηθώ κάθε επιτυχία και στην Ρουμανική Προεδρία. Κυρίε και κύριοι, είχα έρθει εδώ και τον Ιούλιο και τότε είχα πει πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι το αυτονόητο και θα πρέπει καθημερινά να προσπαθούμε να την βελτιώσουμε. Και επειδή είχαμε και δύσκολες συζητήσεις, είχα πει ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα που μας ενώνουν από όσα μας χωρίζουν. Και τα ίδια θα έλεγα και σήμερα. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την πρόκληση της πολύ πολύπλοκης δομής λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχουν όμως παρόλα αυτά πολλά πράγματα που μας ενώνουν ε, και μπορούμε να συνεργαστούμε για να τα λύσουμε. Ώστε δεν υπάρχει καμία εναλλακτική σε αυτήν την συνεργασία και στην διάθεση να βρούμε συμβασμούς. Χαίρομαι για το ότι τους προηγούμενους έξι μήνες ε, καταλήξαμε σε κάποιους συμβιβασμούς και έτσι ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να έκανε κάποια βήματα στην σωστή κατεύθυνση σε πολλά ζητήματα. Δεδομένης της συγκυρίας θα ήθελα να αναφερθώ στο Brexit και τις σχετικές προκλήσεις. Όταν αναλάβαμε την Προεδρία τον Ιούλιο, είχαμε την απέτηση να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την Ευρώπη των 27. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Κομισιόν και τον Μισελ Μπαρνιέ για τις διαπραγματεύσεις, γιατί καταφέραμε και με την δική μας στήριξη να διατηρηθεί η ενότητα των 27 και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να το πούμε και αυτό, δεν ε, μπορεί να κατηγορηθεί για τίποτα στις διαπραγματεύσεις με τη Μεγάλη Βρετανία. Διαπραγματευτήκαμε μια ισορροπημένη πρόταση και διασφαλίσαμε και τις μελλοντικέ μας σχέσεις. Ακόμα και αν είναι αρνητικό το αποτέλεσμα της απόψινής ψηφοφορίας στη Μεγάλη Βρετανία και οι επόμενοι μήνες είναι δύσκολοι, ελπίζω να καταφέρουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι οι 27 και να έχουμε μια κοινή στάση Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν. Η Αυστρία οπωσδήποτε θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει αυτή τη γραμμή. Εκτός από το Brexit έχουμε μια Ευρώπη ε, που εστίασε σε τρία ζητήματα. Πρώτα απ' όλα η ασφάλεια και η καταπολέμηση της παράνομης ε, μετανάστευσης, ε, δεύτερον η εφημερία και τρίτον η γειτονία. Και βεβαίως θα πρέπει να διασφαλίσουμε και την σταθερότητα στη γειτονιά μας. Για το πρώτο θέμα, την ασφάλεια και τη μετανάστευση. Παρά το μπλοκάρισμα που υπήρξε στο θέμα της κατανομής, επετεύχθη κάποια πρόοδο στη συνεργασία με τρίτες χώρες, ειδικά με την Αίγυπτο, αλλά και με άλλες χώρες καταφέραμε να διασφαλίσουμε πως η διάσωση δεν θα γίνεται μόνο από ευρωπαϊκά σκάφη που συνδέεται με ένα άμεσο ειστήριο προς την Ευρώπη, αλλά να υπάρξει διάσωση και από την Αίγυπτο, την Λιβύη και άλλους. Και μετά την διάσωση οι άνθρωποι να επιστρέφουν στη Βόρεια Αφρική. Αυτό οδηγεί στο ότι συνολικά σήμερα έχουμε 95% λιγότερες αφήξεις στην Ευρώπη από το 2015 και το σημαντικό είναι όχι μόνο η μείωση των αφήξεων αλλά και των θανάτων που μειώθηκαν δραματικά σήμερα η κεντρική οδός η μεσογειακή της Ιταλίας de facto έχει κλείσει τις τελευταίες εβδομάδες δεν είχαμε καθόλου αφήξεις καταφέραμε να έχουμε μια συμφωνία των Υπουργών εσωτερικών για την εντολή της Frontex ε, να συνεργάζεται με τρίτες χώρες αλλά να έχει και ένα σημαντικότερο ρόλο και όσον αφορά την ε, ενίσχυσή της με προσωπικό εμείς εξακολουθούμε να στηρίζουμε τις προτάσεις της Κομισιόν και θα ήθελα να ζητήσω και από σας μιλήστε με τους αρχηγούς των κυβερνήσεών σας, με τις κυβερνήσεις σας υπάρχουν κάποιοι που πρέπει να πιστούν όσον αφορά το θέμα της κατανομής. Προσπαθήσαμε να μην επιμείνουμε, αλλά να φέρουμε μία νέα πρόταση. Την υποχρεωτική, αν θέλετε, αλληλεγγύη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τις θετικές της κουβέντες. Για το θέμα της ανταγωνιστικότητας, της ευημερίας, την βιωσιμότητα του οικονομικού χώρου που λέγεται Ευρώπη, ε, δώσαμε βάρος ε, στην βιωσιμότητα της εσωτερικής αγοράς και χαίρομαι για το ότι είχαμε κάποιες ε, θετικές πρόοδους στο θέμα της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς, όπως παραδείγματος χάρη το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον, ετέθη το ζήτημα της φορολόγησης των γιγάντων του διαδικτύου. Έχει υπάρξει μια μεταβολή των απόψεων εντός του Συμβουλίου. Βεβαίως δεν έχουν ληφθεί ακόμα οι αποφάσεις και θα ήθελα και πάλι να σας ζητήσω να μας βοηθήσετε να πείσουμε τις χώρες εκείνες οι οποίες είναι ακόμα επιφυλακτικές για την αηφορία. Ε, αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερος ως Αυστρία και χαίρομαι για το ότι υπήρξε απαγόρευση κάποιων χημικών ουσιών αλλά βεβαίως συμφωνήσαμε και στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τα ΙΟΤΑΧΗ, μια μεγάλη επιτυχία Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιόν. ένα αποτέλεσμα του τριμερούς διαλογού. Η προστασία στο χώρο εργασίας για, από κάποιες ε, καρκινογόνες ουσίας επίσης, ε, ουσίες με και η σχετική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία είναι κάποια βήματα που θα ήθελα να αναφέρω. Μια πραγματικά ισχυρή Ευρώπη, μια ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται και έναν σύγχρονο προϋπολογισμό και ομολογώ πως οι διαπραγματεύσεις ε, αυτές ε, για το ΠΔΠ ξεκίνησαν έτσι ώστε στην αρχή ήμουν πολύ επιφυλακτικός ε, γι' αυτό Είχε δίκιο εδώ ο πρόεδρος της Κομισιόν ότι έπρεπε να μπούμε με ορμή στις διαπραγματεύσεις και τελικά είχαμε μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι ε, περιμέναμε. Και χαίρομαι ε, για το ότι θα ολοκληρωθούν προσεχώς οι σχετικές διαπραγματεύσεις ε, κατόπιν. Έχουμε την πολιτική γειτονίας εκεί ως Αυστριακός βεβαίως ε, είμαι ευγνώμων για το ότι τελικά καταλήξαμε στο να εστιάσουμε σε μια ενίσχυση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Είχαμε μια επίλυση του θέματος ε, του ονόματος ε, και ε, ανοίξαμε κάποια κεφάλαια με την Σερβία και το Μαυροβούνιο, κάτι το οποίο δείχνει πως υπάρχουν πρόπτικες για αυτήν την περιοχή. Και χαίρομαι για το ότι η Ρουμανία και προσεχώς η Βουλγαρία θα δώσουν ιδιαίτερο βάρος στα Δυτικά Βαλκάνια. τον πρόεδρο Ταγιάννη. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το φόρουμ για την Αφρική που είχαμε στην Βιέννη με την Αφρικανική Ένωση όπου προσπαθήσαμε να δούμε τα ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης της Αφρικής και να μην ε, παραδώσουμε αν θέλετε την Ήπειρο αυτή στους Κινέζους κυβερνήσεις ε, είχαν πάρα πολύ καλές επαφές και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους κατέστησαν δυνατό αυτό το φόρουμ. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο αφορά και είναι σημαντικό για εμάς στην Αυστρία ε, για ιστορικούς λόγους, ε, την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του αντισιωνισμού είχαμε κάνει μια διάσκεψη στη Βιέννη με όλες τις εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης ε, και καταλήξαμε και σε συμπεράσματα του Συμβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους ε, τους ε, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων γιατί δεν είναι δυνατόν οι Εβραίοι στα διάφορα κρατημένα να μην αισθάνονται ασφαλείς και πρέπει να το καταπολεμήσουμε αυτό. Τέλος, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν, τον πρόεδρο Γιούνκερ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως ε, τον πρόεδρο, τον κύριο Ταγιάννη, αλλά και τους άλλους αρχηγούς ε, κρατών ε, και κυβερνήσεων για την καλή και επικοδομητική συνεργασία. Προσπαθήσαμε πάντα να κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς για να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταλήξουμε σε συμβασμούς και να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Χαίρομαι για το ότι καταφέραμε κάποια πράγματα σε κάποιους τομείς και δεσμεύουμε ότι ως Αυστρία θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια που υπάρχει κάποιο άρωμα προεκλογικού αγώνα σε όσους θα είναι υποψήφοι τον Μάιο να ευχηθώ καλή επιτυχία και να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Ελπίζω όμως αυτή η συζήτηση να γίνει πάντα με σεβασμό στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης και όπως θέλουν και οι πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία τους έξι αυτούς μήνες και καλή επιτυχία εύχομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you, Chancellor, for your... Σας ευχαριστούμε, Καγκελάρια, για την ομιλία σας, αλλά και για την ε, σαφή ε, δέσμευσή σας και αποσίωση να καταπολεμήσετε τον αντισημιτισμό. Είναι ε, σημαντική προτεραιότητα η ανεξιθρησκεία και ο διαθρησκειακός διάλογος για αυτό το κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά σας, λοιπόν. Σα ευχαριστώ. Και τώρα ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ζαν Κλόντ Γιονκέρ. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σα, μποντζόρνο, κύριε και κύριοι βουλευτέ, κύριε Καγκελάριε, κυρία Υπουργέ και λοιποί. Υπουργοί, κύριε Πρέσβη, Ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας της Αυστριακής Προεδρίας οφείλεται σε εσά. Δεν έχει νόημα να επαναλάβω τα όσα είπε ο Καγκελάριος. Ο απολογισμός της Αυστριακής Προεδρίας είναι εντυπωσιακό, Αν δει κανεί τον αριθμό των συμφωνιών στις οποίες κατέληξαν Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν 134 θέματα είχαν επιτυχή κατάληξη και τα μισά από αυτά με το Συμβούλιο και τα μισά με το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, και συγκρίνω αυτά τα οποία κατάφερε η Αυστριακή Προεδρία με αυτά τα οποία κατάφεραν άλλες προεδρίες ε, από τις οποίες είχαμε μεγαλύτερες απαιτήσεις. Και θεωρώ ότι ο απολογισμός είναι ε, πραγματικά εντυπωσιακό με μια σημαντική εξαίρεση. Εγώ θα ήθελα η Αυστριακή Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να ξεπεράσει αυτήν την αδυναμία στο θέμα του Συμφώνου Μετανάστευσης του ΟΗΕ και να το συνυπογράψει. Ο Σεμπάστιαν το γνωρίζει, του το έχω πει ότι θα ήταν επιθυμητό η Προεδρία του Συμβουλίου να κάνει ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση αντί να στέλνει αρνητικά μηνύματα. Αλλά γεγονός είναι επίσης ότι η Αυστρία δεν είναι η μόνη χώρα που απέριψε αυτό το σύμφωνο. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Αλλά με την εξαίρεση αυτή, όπως είπα αυτή τη στιγμή αδυναμίας, δεν ε, μπορώ πραγματικά να προσάψω τίποτα στην Αυστριακή Προεδρία. Γιατί παρά τις κάποιες ε, προκαταλήψεις ε, που υπήρχαν ε, υπηρέτησε θα έλεγα την ευρωπαϊκή υπόθεση με μεγάλη συνέπεια, ε, συνέχεια και σοβαρότητα. Και πραγματικά απίλαυσα το πώς εμείς ως ε, Κομισιόν είχαμε πάντα απέναντί μας την ετοιμότητα της Αυστριακής ε, Προεδρίας να εγγυηθεί την ενότητα των 27 όσον αφορά τον Brexit, κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ε, η συζήτηση αυτή δεν ήταν μόνο στο επίπεδο των αρχηγών καρτών, αλλά και στο επίπεδο των ειδικών. Εκεί πέρα χάραξε ξεκάθαρες γραμμές η Αυστρία και πραγματικά τη αξίζει κάθε έπαινος. Είμαι ιδιαίτερος ε, ικανοποιημένος ε, για το ότι οθέτησε η Αυστριακή Προεδρία τις προτάσεις μας για την διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων. Εδώ πέρα πρέπει να αναγνωρίσω πως η Κομισιόν βασίστηκε στην πρόταση της αυτή στα όσα είχε προτείνει ο Αυστριακός ε, Καγκελάριος. Τι είχε πει ότι μέχρι το 2000 ένα έτος, θα πρέπει να έχουμε 10.000 ε, άτομα προσωπικό και διαπιστώνουμε τώρα ότι ο Αυστριακός ε, Καγκελάριος και ο Πρόεδρος Κομισιόν ήταν οι μόνοι που επέμεναν σε αυτό το οποίο όλοι ήθελαν και προσπάθησε η Αυστριακή Προεδρία να προωθήσει αυτή και να διατηρήσει ζωντανή αυτή την ιδέα. Παρατηρείτε ότι με ταλαιπωρεί ο λαιμό μου, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι δεν θα με υποστείτε για πολύ. Οπότε θα ήθελα να ξεκαθαρίσω την διγλωσία του Συμβουλίου. Δηλαδή, μα ζητάνε όλοι να κάνουμε κάτι για την προστασία των συνόρων. Κάνουμε κάτι σε συνεργασία με τον Καγκελάριο και μετά έχουμε διάφορες ε, παραπλευρές ε, κινήσεις. Ε, είτε τηρούμε τα συμφωνημένα και αυτά που μα ζητάνε ή καλύτερα να μην μιλάνε κάποιοι. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον ε, καγκελάριο και την Αυστριακή Προεδρία για τη στήριξή τους και σας είπα ότι παρά τις αρχικές επιφυλάξεις ε, που υπήρχαν προωθήθηκε και η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνομιλία στην καγκελαρία και σας είχα παρακινήσει να το προωθήσετε. Το έκανε η Αυστριακή Προεδρία παρά τις επιφυλάξεις που είχε και είμαι ευγνώμων ε, για το ότι επιτέλους μετά την αρχή των τραπεζών έχουμε και μια αρχή ε, για την εργασία. Γιατί είναι λάθος η αίσθηση ότι η Ευρώπη στρέφεται κατά του εργαζόμενου. Όποιος προστατεύει τις τράπεζες πρέπει να προστατεύσει και τους εργαζόμενους και εδώ πέρα μας βοήθησε πολύ η Αυστριακή Προεδρία για το ΠΔΠ, δημοσιονομικές προοπτικές. Πραγματικά και εδώ πέρα οφείλουμε να επενέσουμε και να αναγνωρίσουμε την Αυστριακή Προεδρία. Κατάφερε λοιπόν κάτι το οποίο δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια να πραγματικά φτιάξει έτσι τα διαπραγματευτικά κουτιά όπως ε, λέγονται έτσι ώστε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να έχουν μια διαπραγματευτική βάση που τους επέτρεψε στα θέματα των δημοσιονομικών προοπτικών να επιτύχουν την πρόοδο που χρειάζεται έτσι ώστε τον Οκτώβριο και εδώ πέρα πραγματικά τα κατάφερε η Αυστριακή Προεδρία εγκαίρως να ε, καταλήξουμε κάπου. Οπότε μόνο επένους και εδώ για την Αυστριακή Προεδρία γνωρίζετε πόσο δύσκολα είναι αυτά τα θέματα με τα κουτιά αυτά και τη συναρμολόγησή τους κατάφερε λοιπόν η Αυστριακή Προεδρία να κάνει έτσι τα πράγματα ώστε να προωθηθούν και να σημειωθεί κάποια πρόοδο στις μουσιονομικές προοπτικές. Σας ευχαριστώ και για αυτά τα οποία είπατε για τον αντισημιτισμό δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα φοβόντουσαν οι Εβραίοι συμπολίτε μας να εκδηλώσουν την πίστη τους και η Αυστρία έχει κάποιους ιδιαίτερους λόγους να λέει λόγια σταράτα στο θέμα αυτό ήμουνα και στην Βιέννη από κάποιους μήνες επισκέφθηκα και την εβραϊκή κοινότητα της Βιέννης για να δείξω ότι δεν υπάρχει χώρος ε, για αντισημιτισμό και ρατσισμό στην Ευρώπη. Και στην πράξη νομίζω ε, έδειξε η Αυστριακή Προεδρία ότι θα κάνει